herr präsident αγαπητοί συνάδελφοι κύριε πρόεδρε juncker κύριε πρωθυπουργέ φίτσο για την υπογραφή τη ε, κοινή δήλωση σχετικά με τι νομοθετικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2017. Σα καλοχαιρετίζω. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν για αυτή τη διαδικασία που θα ακολουθείτε με αυτό τον τρόπο οι κοινέ προσπάθειες ε, για του χρόνου να σημειωθούν πρόοδοι σε σχέση με την δήλωση πρόοδοι που πρέπει να επιτευχθούν σε σχέση με την ολοκλήρωση των ε, προγραμμάτων και σχεδίων, σε σχέση με συμφωνία των τριών θεσμικών οργάνων, δεν ήταν καθόλου εύκολο να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Απαιτεί το πολύ βούλη, μεγάλη βούληση για συμβιβασμού από τι τρει πλευρέ. Έδωσε μάχη το Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των εργαζομένων, την καταπολέμηση τη φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή ε, και να ενταχθούν αυτά ως προτεραιότητες στο τέλος, τουλάχιστον από πλευράς κειμένου, καταφέραμε να σημειωθούν πρόοδοι σε αυτά τα θέματα, που πρόοδοι που απαιτούνται να σημειωθούν επιτακτικά. Συγκεκριμένα λοιπόν βήματα και όχι μόνο καινές δηλώσεις ε, κενές περιεχομένου. Πρόκειται συνολικά για την καταπολέμηση και της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και για την βελτίωση της οδηγίας για απόσπαση εργαζομένων που αφορούν άμεσα τα θέματα αυτά τους εργαζομένους μας. Επιτρέψτε μου σε αυτό το θέμα να έχω κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση, ε, που θα αποσαφηνίσω σε σχέση με αυτή τη δήλωση η δήλωση αυτή σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία δεν απεμπολεί καθόλου κάποια θέματα ούτε έγινε βιαστικά και χωρίς ε, δημοκρατικό έλεγχο μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή δεν βιαστήκαμε για να προχωρήσουμε ε, γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι τα όσα δεν έχουν συμπεριληφθεί σε σχέση με αυτή τη δήλωση δεν σταματούν εκεί, το αντίθετο συνεχίζονται Μεγάλο έργο έχει να επιτελεστεί και επιτελείται σε σχέση με νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν νομοθετικά τον έλεγχο και των ε, αρμοδιοτήτων μας όσον αφορά την νομοθεσία. Ο στόχος αυτής της διαθεσμικής διοργανικής συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία έχει στόχο να γίνει η νομοθετική διαδικασία πιο διαφανής και πιο αποτελεσματική. Μια και είναι μέρος λοιπόν αυτό αυτής της δήλωσης, είναι μια συμφωνία για να σημειωθούν συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα, ρεαλιστικά μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό ακριβώς αναμένουν οι πολίτες μας, να δώσουμε χειροπιαστά αποτελέσματα με τις προσπάθειές μας. Και πρέπει λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το μέλημα. Γι' αυτό υπογράφουν οι τρεις πρόεδροι των τριών θεσμικών οργανών, ο κύριος Φίτσο, ο κύριος πρόεδρος Γιούνκερ και εγώ υπογράφουμε αυτή την κοινή δήλωση. Για αυτούς όλους τους λόγους Κυρίες και κύριοι, αποφασίζουμε για ένα σημείο της ημερήσιας διάταξης θεματολογικά που και από τα τρία θεσμικά όργανα, ακόμα και όταν υπογραφεί σήμερα, θα αποτελεί προτεραιότητα εφ' για μας. Κάνουμε ένα τεράστιο βήμα έτσι προς τα εμπρός. Και πρέπει να πούμε ότι και μέσω του Συμβουλίου για πρώτη φορά γίνεται αποδεκτό κάτι τέτοιο. Στόχος και έργο μας είναι λοιπόν αυτή η δήλωση να μπορέσει να ευδοκιμήσει να αποκτήσει σάρκα και οστά. Εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσουμε με αυτό το πνεύμα τη συνεργασία μας με τα θεσμικά όργανα ως Ευρωβουλή, με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικοδομητικά και μετά με τους Προέδρους της Μάλτας και της Εστονίας, θα, Εστονίας να συνεργαστούμε αποτελεσματικά όπως και με τη Σλοβακική Προεδρία κατά τους τελευταίους έξι μήνες. Με ικανοποιεί ιδιαίτερα η ιδιαίτερη, μεγάλη παρουσία των συναδέλφων, ολόκληρους μήνες που συζητούσαν αυτά τα θέματα, δίνοντας ε, σημασία και σπουδαιότητα στα θέματα αυτής της δήλωσης. Ευχαριστώ αυτούς τους συναδέλφους και τους εύχομαι όλα τα καλά και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα λάβει τον λόγο ο πρόεδρος του Συμβουλίου, ο κύριος Φίτσο, παρακαλώ.